και στη συνεργασία Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Φαίνεται πως όχι. Εγκρίνονται οι διορισμοί. Τα πρακτικά θα υποβληθούν την επόμενη εβδομάδα και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα όπως ενεκρίθησαν σήμερα. Διακόπτεται η σύνοδο.